Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Θα γίνει η επίσημη υπογραφή μιας πολύ σημαντικής συμφωνίας μεταξύ Κοινοβουλίου και Κομισιόν. το λεγόμενο μητρό των ομάδων πίεσης Λόμπι. Θα ψηφίσουμε και την έκθεση Κασίνη στην τελευταία σύνοδο του Στρασβούργου. Τώρα θα γίνει η επίσημη υπογραφή. Mm. Είχαμε ψηφίσει στις 10 Μαΐου του 11. Από ό,τι ξέρω το Συμβούλιο θέλει να πει δυο λόγια. Γι' αυτό θα το περιμείνουμε. Την κυρία Υπουργό Μπιούρη να προσέλθει στην αίθουσα για την υπογραφή και καλωσορίζω τους επιτρόπους τον αντι... καθώς και τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής που θα παρίστανται και αυτοί στην επίσημη υπογραφή. Η κυρία Διάννα Γόλης, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι μεταξύ των διαπραγματευτών ήταν η κυρία αντιπρόεδρος Ιζαμπέλ Ντουράν, Ράινερ Βίλαντ επίσης αντιπρόεδρος και ο συνάδελφός μας Κάρλο Κασίνη. πρόεδρος της ΑΦΚΟ. Θα, υπάρχει, θα είναι παρόν και ο εισηγητής, ε, που είναι και ο εισηγητής μάλλον. Παρακαλώ συνάδελφοι, μετά από αυτά που θα μας πει η κυρία Γιούρη που προσέρχεται τώρα, την βλέπω, χαίρετε κυρία Υπουργέ, κυρία Προεδρεύουσα, πριν από την υπογραφή του εγγράφου Τη συμφωνία ε, για το Μητρό των Λόμπι μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής έχετε να πείτε δυο λόγια. Ορίστε κυρία Προεδρεύουσά μου. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας διαβάσω την δήλωση του Συμβουλίου για το Μητρό Διαφάνειας. Το Συμβούλιο θεωρεί τη διαφάνεια ως βασική αρχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνθήκη προβλέπει ότι για να προωθηθεί καλή διακυβέρνηση και να διασφαλιστεί η συμμετοχή και της κοινωνίας ολόκληρης θα γίνεται η εργασία των ομάδων πίσω όσο το δυνατόν διαφανέστερα και όσο πιο κοντύτερα στους πολίτες γίνεται. Γι' αυτό το Συμβούλιο παραμένει δεσμευμένο στην αρχή της διαφάνειας και αναγνωρίζει ότι οι πολίτες αναμένουν όσοι δρούν εξ ονόματός τους στο ενωσιακό επίπεδο αναμένουν υψηλότατα πρότυπα και γι' αυτό καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου να καθορίσουν ένα κοινό μητρό διαφανείας. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι η διαφάνεια πρέπει να οδηγεί τις σχέσεις μας με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και το μητρό αυτό αποτελεί μια σωστή βάση για την διασφάλιση μιας τέτοιας σχέσης διαφάνειας έχει δεχθεί την πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής να συμμετάσχει και αυτό, να συμπογράψει και αυτό το Μητρό. Λυπούμε κυρία Υπουργέ, πρέπει να ζητήσω από τους συναδέλφους, συνάδελφοι, έχει δοθεί ο λόγος στην κυρία Υπουργό, την Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. Σας παρακαλώ λοιπόν να πάψετε τις ιδιωτικές σας συζητήσεις και να ακούτε την κυρία Υπουργό. Συνεχίστε κυρία μου. Ευχαριστώ. Τελειώνω την ανάγνωση αυτή τη δήλωση του Συμβουλίου, λέγοντα ότι το Συμβούλιο δέχτηκε την πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή να συνυπογράψει και αυτό το Μητρό και είναι έτοιμο, διατεθειμένο να παίξει και αυτό ένα ρόλο στον καθορισμό του και είναι διατεθειμένο να συζητήσει τον ακριβή τρόπο με τα δύο άλλα όργανα. Άρα θα έχουμε ένα κοινό μητρό και για τα τρία θεσμικά όργανα. Αυτό θα ήταν άλλωστε και η καλύτερη λύση, να έχουν και τα τρία θεσμικά όργανα ενίο μητρό για εξωτερικά συμφέροντα. Λοιπόν, θα ήθελα και πάλι να σας παρακαλέσω αγαπητοί συνάδελφοι, ε, που σας ανέφερε προηγουμένως τους αντιπροέδρους ε, Wallis Τζιραν Βίλαντ, όπως επίσης και τον πρόεδρο της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Ο εισηγητής κύριος Κάρλο Καζίνη παρακαλείται μαζί με τους αντιπροέδρους που ανέφερα να έλθουν να με πλαισιώσουν στη διαδικασία υπογραφής όπως επίσης και ο πρόεδρο, αντιπρόεδρος συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό Α. Okay.